ψηφοφορίας για έξι ψηφίσματα για την ομοφιλοφιλία. Καταρχάς να κοιτάξουμε το κοινό ψήφισμα έξι ομάδων που θα αντικαταστήσουν τα ψηφίσματα αυτά. Να ψηφίσουμε λοιπόν την παράγραφο 6 του αρχικού κειμένου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε την παράγραφο 8 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορία. Haben alle Dann ist die Abstimmung geschlossen. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Μιλούσαμε για την παράγραφο 8. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε όλοι σας. Εγκρίνεται λοιπόν η ψηφοφορία με 37 ψήφους υπέρ. Να ψηφίσουμε το F τώρα παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το κείμενο. Να ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη παρακαλώ ψηφοφορίας. Μάλε Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Die Resolution ist angenommen mit 60 gegen 60 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε για 7, 7 ψηφίσματα για το Αζερβαϊτζάν για την ελευθερία της έκφρασης και να ψηφίσουμε καταρχάς το ψήφισμα του EFD. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε το κοινό ψήφισμα τώρα έξι πολιτικών ομάδων. Παράγραφος 7. Προφορική τροπολογία της κυρίας Ανδρικάινεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος του ΕΛΚ θα ήθελα να προτείνω τις εξής προφορικές τροπολογίες για την παράγραφο 7. Να αντικαταστήσουμε τις λέξεις deplores the Azerbaijani decision not, δηλαδή αποδοκιμάζουμε την απόφαση της κυβέρνησης να μην, ναι. Να πούμε το εξή στα αγγλικά. Ζητάει από την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν να χρησιμοποιήσουν τις άδειες για τα να ανανεώσουν τις άδειες για τις ραδιοφωνικούς ε, σταθμούς. Υπάρχουν στάσεις για την προφορική αυτή ε, τροπολογία. Όχι. Άρα να ψηφίσουμε την, τροπολο... την, 7, παράγραφο 7 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Υπέρ. Μάλιστα. Κατά. Άποχες. Και το ψήφισμα αυτό λοιπόν εγκρίθηκε. Και έτσι ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες μας. Να σας ανακοινώσω ότι εξ ονόματος ε, Πολωνού ε, δικηγόρου θέλουμε να ζητήθηκε να αρθεί η ασυλία ενός νοδέλφου του Κοινοβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 3 της ε,